Ladies Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από μένα. Έχω την ε, τιμή να προεδρεύω στο πρώτο πάνελ ε, που φέρει τον τίτλο ε, «Τεχνητή νομοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια» και νομίζω ότι μου έκανα αυτή την τιμή γιατί προεδρεύω στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Και αυτή η Επιτροπή ανάμεσα στις αρμοδιότητες της έχει και τις ηθικές, την ηθική διάσταση των νέων τεχνολογιών. Χαίρομαι πάρα πολύ που στο πλαίσιο του διαλόγου με βάση το άρθρο 17 ο Κύριο Σταγιάννη, φιλοξενεί τη σημερινή συνάντηση και η αντιπρόεδρος η κυρία Μαγκίνες και εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Χαρά μου να κηρύξω την έναρξη των εργασιών του πρώτου πάνελ. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο. Σχεδόν κάθε ημέρα ακούμε να λέγονται πολλά για την πρόοδο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη η οποία όλο και περισσότερο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Έχουμε διακεκριμένους ομιλητές και θα ήθελα να τους καλωσορίσω. Έχουμε την κυρία Πρένσακ, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ομάδας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με την ηθική στην επιστήμη και στις νέες τεχνολογίες. Και θα είναι η πρώτη ομιλήτρια. Κατόπιν έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Τάικ, ο οποίος είναι γραμματέας ε, του Συμβουλίου για θέματα πολιτισμού της Αγίας Έδρας. Ακολουθεί ο κύριος Εφραήμ Μύρβης, ε, ο οποίος ε, είναι αρμόδιος για θέματα κοινοπολιτείας ο κύριος Νταμπρόκ, ο οποίος προέρχεται από τη συστηματική θεολογία, πρόεδρος του Ιθικού Συμβουλίου ε, της Γερμανικής Προτεσταντικής Εκκλησίας και τον κύριο Μάικ Φλάντ, ο οποίος ε, ασχολείται με την κριτική ενημέρωση εκ μέρους ε, της Διεθνούς Ανθρωπιστών. Και τέλος έχουμε και την κυρία Μαντιντελβό, που είναι Ευρωβουλευτής, μέλος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και η συγγήτριά μας ε, ε, σχετικά με τους ε, κανόνες, του, τους νόμους του αστικού δικαίου για την ρομποτική η ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοτήνης μπορούν και πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και να εξυπηρετούν την, ε, τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου. Αυτό ήταν το τέλος της παράθεσης ε, από αυτά που έχει πει η Ευρωβουλευτής και επίσης παραθέτω και πάλι όλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται ε, στην αρχή της αυτονομίας και της δικαιοσύνης, στις αρχές και τις αξίες που έχουν κατοχυρωθεί στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο κεφάλαιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η δικαιοσύνη, ε, ισονομία, η κατάργηση των διακρίσεων ε, στην ιδιωτική και στην οικογενειακή ζωή, αλλά ε, και πολλές άλλες αρχές που υπάρχουν στο ενωσιακό δίκαιο, όπως η αποφυγή στιγματισμού, η ατομική ευθύνη, η κοινωνική ευθύνη και η ύπαρξη ηθικών πρακτικών και κωδίκων. Εδώ τελειώνει και η παράθεσή μου. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να συζητήσουμε για το τι ακριβώς σημαίνει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, οποτεδήποτε συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να μην την αμφισβητούμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια κυρία Πράνσακ για να ε, ξεκινήσει ε, με την ομιλία της. Έχετε στη διάθεσή σας 10 ε, λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σφόποντα. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι, είναι τιμή για μένα που συμμετέχω ε, σε αυτή την εκδήλωση και όπως ε, είχα την καλοσύνη να πείτε είμαι ε, πολιτικός επιστήμων, έχω σπουδάσει στη Βιέννη και στο King's College στο Λονδίνο και έχω επίσης την τιμή ε, να μπορώ να σας μιλήσω και για το τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ομάδα ε, για θέματα ηθικής. Πέρα από αυτό όμως ε, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να σας επισημάνω κάποια στοιχεία της ηθικής, της τεχνητής νοημοσύνης που νομίζω αυτή τη στιγμή αξίζουν την προσοχή μας. Ζητώ συγγνώμη που Μερικού από εσά έχω στρέψει την πλάτη μου, αλλά δυστυχώ χρειάζομαι το μικρόφωνο. Και αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και άσκηση τεχνητή νοημοσύνης σήμερα εδώ. Οποτεδήποτε θα σηκώνω το χέρι μου, θα αλλάζει και η διαφάνεια. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτήν την ε, διαφάνεια. Βλέπουμε ότι το περιοδικό ε, Forbes ανέφερε ότι υπάρχει πλέον άνοδος του ρομποτικού εργατικού δυναμικού. Αυτά ανέφερε το περιοδικό. Η τεχνητή νομοσύνη και η ψηφιακή ε, τεχνολογία στην Αγγλία έχουν εισαχθεί στις κλινικές. Ε, ε, βλέπετε ότι εκεί δεν υπάρχει πλέον καθόλου ανθρώπινη παρουσία. Μιλάμε για την διάδοση των ρομπότ. Εδώ βλέπετε ότι είναι το χέρι του ρομπότ και δεν είναι ανθρώπινο το χέρι. Το βλέπετε στη διαφάνεια. Εμείς ως ομάδα ενημερώνουμε για το μέλλον ε, της κοινωνίας. Και βλέπετε εδώ το χέρι είναι ρομποτικό. Ο τρόπος λοιπόν που παρουσιάζουμε τα θέματα ήδη μερικές φορές είναι ένας τρόπος που δείχνει ότι χάνεται η ανθρώπινη διάσταση και δίνουμε προτεραιότητα στην τεχνητή νομοσύνη και στις μηχανές. Και εδώ συμφωνώ με τον Επίτροπο ότι τα κέρια θέματα δεν είναι τα τεχνολογικά. Αυτό που, μάλλον το βασικό ερώτημα είναι τι θέλουμε να είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Ε, να πω το εξής, Όπως όλοι σας γνωρίζετε, ένα από τα πράγματα το οποίο ακόμα και τη συζήτηση, πόσο μάλλον τους κανονισμούς για την τεχνητή νομοσύνη τους καθιστά ιδιαίτερα δύσκολους, είναι γιατί δεν είναι μία πρακτική η οποία χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ενιαίος οικουμενικός ορισμός. Δηλαδή, οι άνθρωποι όταν μιλάνε για την τεχνητή νομοσύνη, δεν μιλάνε όλοι για το ίδιο. Μερικοί, ας πούμε, αναφέρονται στην ε, ε, επιστημονική φαντασία. Και βλέπετε εδώ στην διαφάνεια το τι ακριβώς ε, περιλαμβάνεται στις συζητήσεις για την τεχνητή νομοσύνη. Και ο κατάλογος που δεν είναι, δεν είναι εξαντλητικός. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που εννοούν οι άνθρωποι όταν χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Όμω υπάρχει ένα πράγμα το οποίο ισχύει για όλες τις τις ε, τεχνολογίες ε, κάτω από αυτή την έννοια. Δηλαδή οι τεχνολογίες ε, αφορούν το υλικό και το κοινωνικό στοιχείο, είναι δέσμες κοινωνικές το ίδιο παραδείγματο χάρη και με μια πέτρα. Αν πάρουμε μια πέτρα σε ένα δάσος για να την χτυπήσουμε σε ένα δέντρο και μετά η πέτρα τραπέζι στο έδαφος, αυτή ε, παραμένει ένα στοιχείο της φύσης. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εκείνος που φτιάχνει την τεχνολογία και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να ε, αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως την τεχνολογία στην πράξη. Εδώ λοιπόν και ο Επίτροπος ε, είχε την καλοσύνη ήδη να το επισημάνει. Βλέπουμε το τι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα Ηθικής ε, για την ε, τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τα αυτόνομα συστήματα. Επισημαίνουμε κάποιες αξίες που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές να έχουμε κατά νου οποτεδήποτε διαμορφώνουμε αυτό που θα πρέπει να είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες επ' αυτού, απλά θέλω να επισημάνω το γιατί έχουμε επιλέξει αυτές τις αρχές. Ε, έχουμε μια ειδική σχέση με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δηλαδή τα άτομα δεν τα βλέπουμε σαν ατομιστές που βρέθηκαν στον κόσμο αυτό και είναι ανεξάρτητες οντότητες. Εμείς επισημαίνουμε το ότι τη σχέση αυτή, ε, τη σχέση δηλαδή με την οποία οι άνθρωποι διαμορφώνονται από το τεχνητό περιβάλλον και τα ανάπαλη. Ισχύει και το αντίθετο. Αυτονομία σημαίνει ελεύθερη βούληση, ελεύθερη βούληση των ανθρώπων και ένα πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι σε αυτές τις συζητήσεις είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε την αυτονομία του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μιλάμε για αυτόνομα συστήματα, μιλάμε για αυτόνομα συστήματα όταν μιλάμε για αυτά πάντα σε εισαγωγικά. Η ευθύνη είναι σημαντική διότι συνδέει μάλλον να το πω αλλιώ, μας βγάζει από την αντιπαραγωγική διχοτομία του ατομικού έναντι του συλλογικού συμφέροντος. Το ίδιο ισχύει και για τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την αλληλεγγύη. Δηλαδή, μερικές φορές καλούμεθα να επισημάνουμε αρνητικές πρακτικές που έχουν σχέση με την τεχνητή νομοσύνη. Πρέπει να ε, ε, στυλιτεύσουμε την αδικία. Και αυτό είναι σημαντικό και για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία. Η λογοδοσία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί όσοι λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κακό ε, και τώρα εθελοντικά δημοσιεύουμε τις, τους αλγορίθους μας, η λογοδοσία στην κοινωνία είναι εκείνη η οποία διδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Στις εισαγωγικέ παρατηρήσεις ακούσαμε ότι η διαφάνεια των αλγορίθμων είναι σημαντική, αλλά δεν είναι μόνο αυτό σημαντικό. Σημασία έχει και το τι κάνουν ε, οι αλγόριθμοι, ποιες είναι οι επιπτώσεις τους. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και λογοδοσία για αυτό και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μέσω της νομοθεσίας. Η ασφάλεια, η σωματική ακαιρεότητα, προφανώς αυτά είναι άρρηκτα συνδεμένα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ίδιο και η βιωσιμότητα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να προτρέξουμε, να σκεφτούμε τι σημαίνει η τεχνητή νομοσύνη, η οποία σήμερα ε, δεν ε, λύνει μόνο προβλήματα, αλλά ε, αφορά και μία σειρά άλλων πραγμάτων που θα παίξουν ρόλο στο μέλλον. Και βεβαίως η διαδικαστική αξία ε, όσον αφορά τις διαδικασίες πρέπει να τις σκεφτούμε, ε, να έχουμε μια μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά, ε, γιατί δεν είναι σωστό να λέμε ότι ας αφήσουμε τους ανθρώπους να σκέπτονται και κάτι καλό θα προκύψει. Αν έχει κανείς δει την πολιτική για την ειρήνη στην τελευταία έκδοση του περιοδικού για την επιστήμη. Εκεί οι επιστήμονες είπαν ότι οι πολίτες, το κοινό μπορεί να καταλήξει σε πολύ καλές λύσεις. Τελειώνοντας, θέλω πολύ σύντομα να επισημάνω τρία θέματα ε, που πρέπει να έχουμε κατά νου ε, πέρα από όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στην ομάδα ηθικής. Ας ε, έχουμε κατά νου την πολιτική οικονομία μέσα στην οποία δημιουργείται η τεχνητή νοημοσύνη. Μερικοί και εγώ ισχυριζόμαστε ότι ένα από τα αίτια που υπάρχουν μονοπόλια και που τα μονοπόλια γίνονται ο νέος Λεβαθιάν, δηλαδή γίνονται κάτι που ο που προκύπτει, που φαίνονται, αλλά που τελικά αποκαλύπτουν ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ε, όσον αφορά την ε, ανθρώπινη κοινωνία, τον έχουμε ένα νέο Λεβαθιάν. Αυτό ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει να σκεφτούμε ε, ποιες τι είδου ρυθμίσεις θεσμικές και άλλες χρειαζόμαστε. Και εδώ χρειαζόμαστε και την πολιτική κατανόηση της ηθικής. Τι εννοώ, δεν εννοώ το κομματικό πολιτικό της ηθικής όπου συζητάμε ε, για τις θέσεις ε, των κομμάτων ή για διάφορες θρησκευτικέ απόψεις. Εγώ εννοώ πολιτική ηθική που πραγματικά προσπαθεί να εξετάσει την καλή ζωή, την καλή κοινωνία και στυλιτεύει ε, τις ε, αδικίες ε, οπουδήποτε αυτές προκύπτουν. Επίσης θέλω να πω ότι κατά την ψηφιακή εποχή, την εποχή των big data και της τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορούμε πια να έχουμε κατά νου ότι θα τα καταφέρουμε μειώνοντας τους κινδύνους. Ε, χρειαζόμαστε πολύ καλύτερους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ζημιάς, που η ζημιά θα προκύψει από την ε, νομοθετημένη χρήση ε, των δεδομένων. Το βιβλίο που βλέπετε εδώ που σας προβάλλω στη διαφάνεια, βλέπετε ότι σίγουρα από τα δεδομένα θα προκύψουν ζημιές. Να σε επισημάνω ένα συνάδελφο, το Λίλο Χάγκεντοφ, ε, που ε, δημοσίευσε αυτό το βιβλίο την προηγούμενη εβδομάδα, όπου εξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ηθική και καταλήγει στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπησέρχεται σε, και παίζει ρόλο σε πολλά από τα τελευταία σκάνδαλα. Υπογραμμίζει ότι η επιστήμη και οι κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη υποφέρουν. Εκείνος λέει ότι χρειαζόμαστε, ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα με ηθική και δεν χρειαζόμαστε κανόνες. Με αυτά κλείνω την ομιλία μου και προσβλέπω στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, στον οποίο θα ήθελα να δώσω το λόγο, είναι ο Πολ Τάιγκ, αρχιεπίσκοπος από το Συμβούλιο Πολιτισμού των Καθολικών, της Καθολικής Εκκλησίας. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε. Τα σχόλια που θα κάνω είναι, προκύπτουν από κάποιες σχέσεις, ε, σκέψεις μάλλον που προέρχονται από την καθολική παράδοση, χωρίς να υπάρχει κάποιο συμπέρασμα ή κάποιο δόγμα είναι απλώς κάποιες πρώτες σκέψεις που έχουν τη σημασία τους όμως. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο της ομάδας ψηλού επίπεδου. Πάνω απ' όλα εδώ προσπαθούμε να πυροδοτήσουμε τη δημόσια συζήτηση, τη δημόσια διαβούλευση που είναι κρίσιμη αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, είναι σαφές ότι υπάρχει μια δέσμευση ε, σε αυτή τη συζήτηση ε, να μην αποκλείσει κανέναν υπάρχει μια μεθοδολογία. Προσπαθούμε να βρούμε μια γλώσσα, μια ορολογία ε, που να είναι συνεπής, το οποίο δεν είναι πάντα προφανές. Δίνεται επίσης ε, έμφαση στην ηθική, ε, χωρίς να φτάνουμε σε συμπεράσματα βιαστικά. Το κριτήριο του, το ανθρωποκεντρικό επίσης είναι εξαιρετικό. Είναι, πάει προς την κατεύθυνση. Επίσης η δέσμευση του ε, υπάρχει ένας μηχανισμός αξιολόγησης ε, είναι επίσης σημαντικό. Να πω δύο, τρία πράγματα από ηθικής πλευράς. Ορισμένες φορές ε, προσπαθώ να καταλάβω τι εννοούμε όταν μιλάμε για ηθική. Τι σημαίνει, τι είναι καλό και τι είναι κακό και πώς καθορίζουμε το καλό και το κακό. Ορισμένες φορές η χρήση της ηθικής συχνά έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο, πώς θα ακολουθήσει τις ιδέες μας, ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή να χειραγωγηθεί το θέμα της ηθικής. Δεν μπορούμε όμως να, να περιορίζουμε την ηθική σε, τέτοιου υπολογισμού. υπολογισμούς. Πρέπει να προσπαθήσουμε η ηθική να, να μας οδηγήσει να κάνουμε το καλό, ακόμα και αν αυτό έχει ένα κόστος. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε περισσότερο για την συνείδηση της προσωπικής ευθύνης των ανθρώπων, ε, να πάρουν αποφάσεις ε, που δεν είναι απλά ηθικές αποφάσεις με τη στενή έννοια, αλλά που καθορίζουν το ποιοι είμαστε και το ποια κοινωνία θέλουμε να φτιάξουμε. Η σημασία λοιπόν των προσώπων, των ατόμων που παίρνουν θέση και κάνουν συγκεκριμένε επιλογές. Διότι ορισμένε φορές ε, μιλάμε για τους μηχανικούς, μιλάμε για την τεχνολογία που, που δεν δέχτηκαν να κάνουν κάποια πράγματα ε, λόγω της θέση των χωρών τους. Λοιπόν, ανοίγουν και κάποιες πιο βαθιές συζητήσεις. Αν θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα ε, αυτήν την ανθρωποκεντρική φύση, ε, πρέπει να σκεφτούμε τι είδους ζωή θέλουμε να φτιάξουμε, τι είδους κοινωνία θέλουμε να φτιάξουμε. Ποιο είναι το όραμά μας τελικά, προς τα που πάμε. Τι είναι αυτό που θα προωθήσει πραγματικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ε, είναι πολύ σημαντική και η συζήτηση ε, για τα δικαιώματα αλλά πρέπει να καταλάβουμε πώς αντιλαμβανόμαστε τα δικαιώματα. Ε, διότι για μας, ε, στην κουλτούρα μας, στην παράδοσή μας, ε, τα δικαιώματα αυτά είναι αυτα, αυταπόδεικτα, είναι, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Επίσης, τι σημαίνει το να είμαστε κοινωνικά όντα. Ζούμε σε κοινότητες, σε κοινωνίες. Χρειαζόμαστε οι τους δε. Δεν είμαστε απλά άνθρωποι που θέλουμε να έχουμε μια συναλλαγή ή ένα συμβόλαιο στα πλαίσια της κοινότητας. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή αξιοπρέπεια. Ο, ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε, παραδείγματο χάρη, στην αξιοπρέπεια της οικογένειας. Στο κοινό σπίτι που μοιραζόμαστε όλοι πρέπει να το καταλάβουμε αυτά τα ζητήματα. Τέλος, ε, να πω δύο-τρία ακόμα πράγματα. Ε, θα το πω γιατί είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να υπογραμμίσουμε και το κάνουμε εμείς στην παραδοσή μας. Ε, το το πόσο καλή είναι η, η, η, η επιστήμη και η τεχνολογία. Το να μάθουμε, που μα βοηθάει να καταλάβουμε περισσότερα για εμά, για τον κόσμο, να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση αυτή για το καλό τη ανθρωπότητα. Αυτό είναι ευλογία. Είναι κάτι θετικό και πρέπει πάντα να το ε, γνωρίζουμε αυτό και να το αναγνωρίζουμε. Ε, είπε ο επίτροπο νωρίτερα ότι οι τεχνολογικέ δυνατότητε έχουν ξεπεράσει τι ηθικές δυνατότητε. Ε, Ορισμένε φορές ε, μιλάμε για διπλή χρήση, διτή χρήση. Ε, σκεφτόμαστε πολύ συχνά το τεχνολογικό πρέπει, ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα από τεχνολογικής πλευράς. Ο Πάπας Φραγκίσκος για το περιβάλλον έχει πει κάποια πράγματα. Ε, υπάρχει ένα τεχνολογικό τεχνοκρατικό παράδειγμα. Πολλά τεχνολογικά προϊόντα παράγονται ε, σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό, οικονομικό, πολιτιστικό περιβάλλον με συγκεκριμένες προτεραιότητες που προϋπάρχουν. Το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο ο κόσμος μας ήδη σημαδεύεται από μεγάλες ε, ανισότητες, μεγάλη έλλειψη δικαιοσύνη. Μήπω υπάρχει τελικά ο κίνδυνο ότι η παραγωγή τη τεχνητή νοημοσύνη που θα ε, δημιουργήσει πολύ μεγάλα εμπορικά πλεονεκτήματα και εξουσία για λίγους και όλο και λιγότερους τελικά. Αυτό λοιπόν θα είναι προς το καλό των, του συνόλου της ανθρωπότητας. Υπάρχει η ανισότητα η οικονομική, η ηλική, αλλά και υπάρχει, η ανισότητα ε, η δημοκρατική. Ποιος μπορεί να επηρεάσει περισσότερο την εξουσία, ποιος μπορεί να ελέγξει, πού λογοδοτούν αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει. Είναι και αυτό που δημιουργεί ρογμέ στην ενότητα των, ανθρώπων. Πολύ σημαντικό το θέμα λοιπόν από νομοθετική πλευρά, από ηθική πλευρά, αλλά υπάρχει και θέμα ευαισθητοποίηση των ανθρώπων και των επιλογών του. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Thank you as well. Ευχαριστώ πολύ να ακούσουμε τώρα τον Εφραίμ Μυρβής, ε, τον ε, αρχιραβίνο ε, των ε, ενωριών του Commonwealth. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργάνωσε αυτή τη διάσκεψη εδώ σήμερα. Είναι χαρά μου να συνεισφέρω κι εγώ με κάποιες σκέψεις από εβραϊκής πλευράς. Στην Πράγα του 16ου αιώνα, το, ο περίφημος Ραβίνος, ο Μαχαρέλ, σύμφωνα ε, με τα λεγόμενα, δημιούργησε τον Γκόλεμ. Το Γκόλεμ ήταν ένα είδους ρομπότ, μια εικόνα, που, είχε φτιαχτεί από ε, λάσπη και τον Γκόλεμ πήρε ζωή. Δίνουν, επειδή του έδωσε το όνομα ο Ραβίνος. Το, δημιούργησε αυτό ο Ραβίνος για να ενισχύσει τη ζωή, να δημιουργήσει ζωή. Μετά από λίγο καιρό όμως τον το Γκόλεμ είχε πια δικό του εγκέφαλο και βγήκε εκτός ελέγχου και άρχισε να είναι ε, επικίνδυνο για την κοινωνία, για τη ζωή. Αυτή η ιστορία είναι πριν από 500 χρόνια, έτσι. Μας στέλνει όμως ένα μήνυμα για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίω, εμεί καλωσορίζουμε τον εξχρονισμό, την πρόοδο, την τεχνολογική, που με τόσο εκπληκτικό πράγμα, με τόσο εκπληκτικό τρόπο μάλλον ενισχύει και βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά υπάρχουν και σημαντικά αρνητικά στοιχεία. Ποιο είναι το πιο σημαντικό σημείο της βίβλου. Γέννηση κεφάλαιο 5.1. Ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' και, ο ομοίωσή του. Δείχνει λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν φτιαχτεί κατ' ομοίωση και του Θεού, οπότε όλοι οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι ιεροί. Και περιγράφει αυτό και την τον ανθρωπισμό μας έχουμε την εικόνα του Θεού και χάρη στην ψυχή μας μπορούμε με την ελεύθερη βούληση να κάνουμε ηθικές κρίσεις. Και αυτή η δυνατότητα να κάνουμε μια ηθική κρίση είναι που μας καθορίζει ως ανθρώπους. Στην έξοδο μας λένε ότι οι Ισραηλίτες δημιούργησαν ένα ε, ναό για το Θεό περιγράφουμε τους χάχαμλεβ εκεί, μια λέξη που νομίζω δεν υπάρχει σε άλλες ε, γλώσσες, που είναι καλόκαρδοι και σοφοί άνθρωποι. Είναι και τα δύο μαζί, όλες οι αρετές ε, του ανθρώπου. Αυτοί λοιπόν που δημιουργούν τον ναό του Θεού, που δημιουργούν και το μέλλον της ανθρωπότητας, πρέπει να βρουν αυτήν την το ιδανικό μείγμα της σκέψης και των συναισθημάτων. Συναισθημάτων που προέρχονται από μια ψυχή. Τώρα ένα μηχάνημα μπορεί να έχει σκέψεις από αυτούς που το προγραμματίζουν. Αλλά δεν έχει καρδιά. Δεν έχει ψυχή. Δεν μπορεί να υπάρξει ως όν με συναισθήματα. Οπότε δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο από μία μηχανή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κάθε μέρα οι Εβραίοι που γνωρίζουν πρέπει να συνδυάζουν το μυαλό και την καρδιά για να είναι πραγματικοί άνθρωποι. Ο κίνητος με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι εγκαταλείπουμε την ηθική μας, τις ηθικές μας αξίες και τις εγκαταλείπουμε στα χέρια αυτών των μηχανών αν έχουμε ένα αυτοκίνητο χωρίς ε, οδηγό, κάτι που θα συμβεί στο μέλλον από ό,τι φαίνεται για όλους μας, και αν αυτό το αυτοκίνητο απλά ε, ετοιμάζεται να, να έχει ένα δυστύχημα και πρέπει να γίνει μια επιλογή, να υπάρχει μια ηλικιωμένη γυναίκα αριστερά και ένα παιδάκι δεξιά, τι θα κάνει λοιπόν το αυτοκίνητο τότε, ε, ε θα προστατεύσει τη ζωή του επιβάτη, του ηλικιωμένου, του παιδιού, θα το αποφασίσει αυτό ένα μηχάνημα. Ε, θα μου πείτε όχι. Οι άνθρωποι οι οποίοι προγραμμάτισαν ε, το, το μηχάνημα αυτό έχουν την ηθική, έχουν κάνει τις ηθικές επιλογές αυτές. Έχουν ένα ηθικό κώδικα. Όμως αυτό γίνεται σε επίπεδο επιχειρήσεων. Μιλάμε για επιχειρήσεις και δυτικά συμβούλια επιχειρήσεων που έχουν ορίσει τους ανθρώπους αυτούς και βάσει, βάσει ποιων κριτηρίων παίρνουν οι αυτές και σε ποιον λογοδοτούν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό, πέρα από τη στρατηγική σημασία ε, της σημερινής συζήτηση μαζί με τόσε άλλε συζητήσει που θα γίνουν, να δώσουμε μεγαλύτερη ένταση σε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να ακουστεί περισσότερο αυτό το θέμα, να είμαστε πιο ανοιχτοί, να λογοδοτούμε, να είμαστε πιο διαφανείς πρέπει να γίνει κατανοητό πόσο κρίσιμο είναι για το μέλλον τη ανθρωπότητα, διότι περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι που διακυβεύεται, να θέσουμε κάποια όρια, να έχουμε κάποιες τι γραμμέ. Πρέπει ε, τα καλύτερα μυαλά, ε, πολιτικοί ηθήνοντε, θρησκευτικοί ηθήνοντε, επιστήμονε που να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή. Και χρειάζεται ρύθμιση τώρα, να μάθουμε από τα παραδείγματα και από τα λάθη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Τώρα, τώρα προσπαθούμε να καλύψουμε εκεί τα κενά σε κάποιο βαθμό τα, τα κοινωνικά δίκτυα, δίκτυα μέσα δικτύωση μα ξέφυγαν. Ξέφυγαν από τον έλεγχο. Εδώ όμω με την τεχνητή νοημοσύνη προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε να έχουμε την κατάλληλη ρύθμιση για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τι εξελίξει και να τι ελέγξουμε. Και εμεί έτσι να κάνουμε το πιο σωστό, το πιο υπεύθυνο, να είμαστε εμεί αυτοί που ελέγχουμε το τι συμβαίνει και όχι το αντίθετο. Όταν δημιούργησε τον άνθρωπο ο Θεός, του είπε ότι έχει δύο ευθύνες. Να εργαστεί στον κόσμο αυτόν και να τον διαφυλάξει. Και τα πάμε αρκετά καλά για το πρώτο, για την εργασία. Εργαζόμαστε στον κόσμο. Δημιουργούμε. Είμαστε παραγωγικοί. Ήρθε η ώρα όμως να αριστεύσουμε και σε ό,τι αφορά το δεύτερο που μας ζήτησε ο Θεός. Να διαφυλάξουμε τον κόσμο αυτό πριν είναι πολύ αργά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πίτερ Ντάμπροκ, ο οποίος είναι καθηγητής συστηματικής θεολογίας, για έξι λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Εγώ θα ασχοληθώ με την τεχνητή νομοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η έκφραση της ελευθερίας ε, και αυτοδιάθεση είναι βασικά χαρακτηριστικά. Κανείς όμως δεν ασχολείται με την αξιοπρέπεια. Βέβαια, έχουμε πολλές ε, θρησκευτικέ ε, ομολογίες οι οποίες θεωρούν ότι θα μπορούσαν αυτό να το αγνοήσουν. Αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ελευθερία και η αυτοδιάθεση, η, ε, το εύθραυστο στοιχείο που αφορά όλους τους ανθρώπους ε, και η εξάρτηση των ανθρώπων από την κοινωνία και από την εύρυθμα λειτουργούσα κοινωνία. Όταν πρόκειται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ε, που αμφισβητείται από την τεχνητή νομοσύνη, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πολλές βελτιώσεις ε, που προσφέρει, τις υποσχέσεις, ε, αυτά που εμείς ως κοινωνίες και ως άτομα δεν έχουμε μόνο ως ευθύνη για να δράσουμε, αλλά οφείλουμε και να απέχουμε από παράλογες πράξεις. Από την άλλη πρέπει να έχουμε κατά νου ε, την ε, διαλυτική τάση ε, που είχε η τεχνολογία και η τεχνητή νομοσύνη στο σύνολο της διαβίωσής μας και στις κοινωνίες μας. Όσον αφορά τις επιπτώσεις της τεχνητής νομοσύνης, κάνω ρητορικές ερωτήσεις. Πώς ακριβώς θέλουμε να υπερασπιστούμε την ειρήνη και την αυτοδιάθεση τη στιγμή που εμείς ως άτομα και ως ομάδες μπορούμε και γίνουμε γινόμαστε όλο και περισσότερο αντικείμενα μιας ε, ισχυρής τεχνολογίας ελέγχου και πώς είναι δυνατόν ε, προσωπικά και κοινωνικά να αντισταθούμε όταν ε, βλέπουμε ότι και εμείς ε, γινόμαστε έρμεα εκείνων που προσφέρουν ευχάριστες λύσεις σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Τα περισσότερα από όλα αυτά συμβαίνουν παρότι επηρεάζονται ομάδες ατόμων και μεμονωμένα άτομα και όλο και περισσότερο οι προγραμματιστές δεν κατανοούν τη λογική που διέπει τη λήψη αποφάσεων ή ε, τους αλγόριθμους. Πώς μπορούμε λοιπόν να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την ε, διαλυτική τεχνολογία για να μην χάσει ο άνθρωπος την κυριαρχία στην τεχνολογία, για να μπορούμε να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επ' αυτού θα εκφράσω τρεις σύντομες απόψεις. Πρώτον, έχουν, έχει ασκηθεί κριτική και έχουν πει, υποθεί πολλά ε, για την αξιοπιστία της τεχνητής νομοσύνης και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να αφαιρθώ κυρίως στα θαυμάσια ε, σχόλια της ε, Προτεσταντικής Εκκλησίας της Γερμανίας που μπορείτε να βρείτε στο φάκελό σας. Παρ' αυτά, εγώ συμφωνώ και με την προσέγγιση ε, αυτής της ε, ομιλίας ε, που θεωρώ ότι είναι καινοτόμος με την έννοια ότι για πρώτη φορά διαφοροποιείται και κατά δεύτερον εξισορροπεί το σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συναφή και δεύτερον εντοπίζονται τα τεχνικά μέσα και τρίτον επιβεβαιώνεται η κριτική προσέγγιση των προϋποθέσεων. Δεύτερον, αυτό έχει και ακόμα μεγαλύτερη σημασία, για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ανθρώπινη αξιοπρέπεια την εποχή της τεχνητής νομοσύνης, οφείλουμε να επανεφεύρουμε την προστασία των δεδομένων. Για το Γερμανικό Συμβούλιο Ηθικής, του οποίου προείσταμε, είναι απόλυτα σαφές ότι η κλασική προσέγγιση της προστασίας των δεδομένων που εξακολουθεί να επηρεάζει το GDPR, ε, παρότι έχει τεθεί πλήρω σε εφαρμογή, δυστυχώ είναι ξεπερασμένη αυτή η εκδοχή. Για να μπορέσουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε την αυτοδιάθεση, οφείλουμε να έχουμε μία αλλαγή, η οποία αποτελείται να περάσουμε από, μία, από ένα παραδοσιακό προσανατολισμό της ε, ξεπερασμένη μεθόδου για την προστασία των ενδομένων, να περάσουμε ίσω σε μία άλλη ε, προσέγγιση, η οποία είναι πιο ανοιχτή με την έννοια ότι εκεί θα ενταχθούν πάρα πολλές ε, διαστάσεις που αφορούν στην κυριαρχία των δεδομένων, δηλαδή ε, μια πραγματική ενημερωτική αυτοδιάθεση. Αυτό το data sovereignty, η κυριαρχία των δεδομένων, προσφέρει όλα τα τεχνικά μέσα για να μπορούμε να διαφυλάξουμε τα δεδομένα που προέρχονται κυρίως από το αντικείμενο. Και μετά πρέπει να δεχτούμε την επιτάχυνση της ε, τεχνολογίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια ευημερούσα ζωή κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Για να τα καταφέρουμε αυτά ε, δεν χρειάζεται μόνο να ε, προάγουμε τις δεξιότητες, αλλά να προάγουμε την κλασική βιβλιογραφία περισσότερο από ποτέ έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα 4C, Communication, Collaboration, Creativity και Critical Thinking. Και γι' αυτό λοιπόν συστήνω να διαβάσουμε διαβάσετε κλασικά κείμενα όπως ε, τη βίβλο, τον Σέξπιρ, ε, βιβλία μαθηματικής, ξένες γλώσσες, να ασχοληθείτε με τη μουσική και τέλος να ασχοληθείτε και με τον αθλητισμό. Νομίζω ότι αυτά χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Ε, και δεν θα ήμουν θεολόγος αν δεν ήμουν ακράδαντα πεπισμένος ότι οι θρησκευτικέ παραδόσεις μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, τα θεμέλια της συνύπαρξής μας την εποχή της τεχνητής νομοσύνης προσφέροντας πλατφόρμες πέρα από την οικονομία των πλατφορμών για το κοινό καλό και σπάζοντας ε, την τεχνητή νοημοσύνη ε, σε ε, διάφορα τμήματα. Αυτό είναι επίγον και νομίζω ότι αυτό στηρίζει και την παράδοση και βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης give Mr. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Μάικ Flood, ο οποίος ε, εκπροσωπεί Critical Information της ε, Διεθνής των Ανθρωπιστών. Για 6 λεπτά, παρακαλώ. Κύριε uh, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω, να επαναλάβω αυτά που είπε και ο πρόλαλή σα, δηλαδή ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή τη συνάντηση που βοηθάει να υπάρχει και συμμετοχή του κοινού σε αυτό το πόσο σημαντικό θέμα. Ο ουμανισμός είναι μια θετική προσέγγιση στη ζωή που βασίζεται στην επιστήμη και στην ε, ανθρωπότητα. Ο ουμανισμός επιβεβαιώνει τη λέξη αυτονομία και τη λέξη αυτονομία του ατόμου και προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία που είναι συμβατή με τα δικαιώματα των άλλων. Και θα ήθελα να αναφέρω κάτι και να αναφέρω και τρεις ανησυχίε μου. Αυτό που θέλω να πω αφορά τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, παραπληροφόρηση, αυτά ε, προάγονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα οι θεωρίες ε, περί ε, σκευωρίας έχουν επεκταθεί ε, λάθος πληροφορίες ε, που έχουν ως στόχο να εξοργήσουν. Αυτά διαδίδονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής, κοινωνικής δικτύωσης και ζημιώνουν την ανθρώπινη ζωή. Ε, σε πολλές περιπτώσεις βοηθούν και να αναπολώσουν συζητήσεις και υπονομεύουν τη δημοκρατία. Υπάρχει μια ειδική μονάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κάθε μέρα ασχολείται με αυτά ε, τα μέσα κοινωνικής διοίκησης, γιατί, κοινωνικής δικτύωσης, γιατί εντοπίζει κάποιες ιστορίες οι οποίες μπορούν να έχουν και πολιτικές επιπτώσεις. Ε, οι διάφορες φήμες για απαγωγές παιδιών διαδίδουν γίνονται μέσα από το WhatsApp, αυτά στην Ινδία, αλλά και αλλού στην Μιανμάρ επίσης καταδικάστηκε ο ρόλος του Facebook από τα Ηνωμένα Έθνη. Μπορούμε να περιμένουμε και χερότερα τη στιγμή που εμφανίζονται βίντεο ε, στο YouTube, στο Instagram και στο Twitter και βρισκόμαστε σε ένα κόσμο όπου τίποτα από αυτά που ακούμε εδώ δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Η τεχνολογία ήδη υπάρχει και τουλάχιστον ένας φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου ε, προβλέπει ότι φέτος θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός με βάση ε, ψεύτικες, ε, διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αυτό λοιπόν που με ανησυχεί είναι ότι θα ήταν προς όφελος ε, των επιχειρηματιών να επηρεάσουν τα μέσα ενημέρωση με έναν τρόπο που δεν είναι ε, ευκταίος. Κάποια στελέχη χρησιμοποιούν όρους όπως ε, humanism και humanistics για να προάγουν τη δουλειά τους. Και εγώ ως ανθρωπιστής αυτές τις λέξεις τις βρίσκω αρνητικές και παραπλανητικές. Τα τελευταία χρόνια η Google και η Amazon έχουν διασφαλίσει πολλά μοντέλα που έχουν με τα συστημικά προϊόντα έχουν μία μέθοδο να βγάζουν κάποιες λέξεις, να τις επιλέγουν, μετά να κάνουν διαφήμιση με βάση αυτές τις λέξεις και αυτά να έχουν σχέση ε, με το ε, υπόβαθρο και με την προέλευση των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έχει σχέση με το σκληρό καπιταλισμό. Η τεχνολογία των μεγάλων εταιριών μας έχει προσφέρει πάρα πολλά. Τώρα όμως ε, θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την ιδιωτική σφαίρα και αυτά είναι μόνο η αρχή, η ευφύης πόλης, ε, το ίντερνετ των πραγμάτων. Ε, όλα αυτά βρίσκονται ε, στην παιδική του ηλικία αυτή τη στιγμή. βλέπουμε λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί με τρόπους που να μπορούν να την κατανοήσουν ακόμα και οι σχεδιαστές της και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αθέλητες συνέπειες. Γι' αυτό θεωρώ ότι η κοινωνία πρέπει να επιμείνει οι σχεδιαστές τεχνητής νοημοσύνης να σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, πριν ε, πάρουν άδεια ε, χρήσης των, σχεδίων τους. Εξαρτώμετα από την τεχνολογία, από τους αλγορίθμους, αυτή αντικαθιστούν όλο και περισσότερο τη λήψη αποφάσεων. Το βλέπουμε με το Google Searching, με την Amazon, με αυτόματες αναλύσεις ε, για οικονομικά στοιχεία και διάφορα άλλα που διαδίδονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά ενθαρρύνουν πολλούς ε, το να ανεβάζουν στοιχεία που γίνονται viral. Ε, πέρυσι η Google καταδικάστηκε γιατί έδειξε ένα ρομπότ που μίλαζε, μίλαγε τόσο φυσικά που πολλοί πίστευαν ότι ήταν άνθρωπος. Αυτό μπορεί να είναι ε, έξυπνο, αλλά δεν σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και τι γίνεται και με την τεχνολογία αναγνώρισης του ατόμου. Ίσως ε, όταν ε, ελέγχονται τα διαβατήρια ή όταν κάνει κανείς σκάνερ σε φυλακισμένους, αλλά τι γίνεται σε απλή χρήση. Και το τρίτον, πρέπει να αποφασίσουμε μέχρι πού θέλουμε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε τις ατέλειτες συνέπειες. Η εκμάθηση με μηχανές χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη, στην ιατρική, στα οικονομικά και έτσι ε, προκύπτουν δύσκολες ερωτήσεις ε, του να μεταφράζονται γενικές ηθικές αρχές ε, σε πρακτικές που να είναι οικουμενικά κατανοητές. Νομίζω η κοινωνία των πολιτών πρέπει να επιμείνει έτσι ώστε να υπάρχουν κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη που δεν θα σέβονται μόνο την ιδιωτικότητά μας ε, αλλά επίσης θα είναι και όλα αυτά ε, διαφανή, θα υπάρχει απόλυτη λογοδοσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τέλος η κυρία Μάντι Ντελβό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια ε, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για τη ρομποτική. Έχετε μόλις 5 λεπτά γιατί είστε και εντός έδρας. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη διότι υποτίθεται ότι εγώ θα κάνω και τα συμπεράσματα αυτής της ε, ενδιαφέρουσα αλλαγή ε, απόψεων. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα. Δεν θα συνοψίσω αυτά που είπε ο Επίτροπος βέβαια. Αν μου το επιτρέπετε όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπράισακ που είπε ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο ηθικές αρχές αλλά και νόμους διότι οι ηθικές αρχές καλές είναι βεβαίω. αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Και θέλω βεβαίω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας θεωρώ δεδομένο ότι όλοι θέλουμε να γίνει μια πραγματική συζήτηση για το ποιο είναι ο τελικό μα στόχο σε ό,τι αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι απλώ κάποιε όμορφε και έξυπνε συσκευέ. Και θέλω να παραθέσω εδώ αυτό που είπε ο επίτροπο, να γίνουμε καλύτεροι πολίτε και καλύτεροι επαγγελματίε. Ε, πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική αυτή η προσέγγιση. Δεν θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τη δική μα νοημοσύνη. Είναι ένα εργαλείο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για το καλό της ανθρωπότητας. Να υπογραμμίσω βεβαίως ότι όλοι τονίσατε ότι η ηθική δεν είναι απλά ένα επιχείρημα, ένα εμπορικό επιχείρημα ε, που πουλάει δηλαδή. Είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με την, την ίδια την φύση του ανθρώπου και του, του τι θέλουμε να κάνουμε ως κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η συζήτηση Θέλουμε λιγότερες ανισότητες. Νομίζω συμφωνούμε από αυτού, ε, έτσι ελπίζω. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχει κίνδυνος νομοσύνη να αυξήσει τις ανισότητες. Κάποιοι από εσά είπαν πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Σε ό,τι αφορά το τι διακυβεύεται. Και να μην μπαίνουμε στον πειρασμό όλων αυτών των όμορφων πραγμάτων που μας προσφέρει η τεχνητή νομοσύνη θα είναι δύσκολο να αντισταθούμε. Θέλω τώρα να αναφερθώ σε δύο στοιχεία που ακούστηκαν ξανά και ξανά. Διαφάνεια. Θέλουμε όλοι να ξέρουμε τι συμβαίνει στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν αρκεί όμως η διαφάνεια. Χρειάζεται και λογοδοσία. Αυτοί που σχεδιάζουν, που δημιουργούν τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να λογοδοτήσουν στην κοινωνία και εμεί ω κοινωνία των πολιτών αλλά και ω πολιτικοί θύνοντες θα πρέπει να δούμε ε, σε ποιον λογοδοτούν αυτοί που δημιουργούν τα προγράμματα. Αυτό είναι το πιο επίγον νομίζω. Μπορούμε τώρα να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει χρόνος θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πραγματική συζήτηση από όλου και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Ο ανθρωπισμός ε, ήταν στο κέντρο όλων των παρεμβάσεων. Μιλήσαμε για τροποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ελέγχθη ε, ε να αποφύγουμε επιπτώσεις που δεν επιθυμούμε κάποια από αυτά τα υπέροχα εργαλεία δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στην τρέλα. Αυτά. Προσπάθησα να συνοψίσω τις, την εντύπωση που αποκόμισα από τις συνεισφορές σας και ελπίζω και πιστεύω ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν καθετές γραμμές για το έργο μας ως πολιτικούς θύνοντες, ως νομοθέτες αλλά και συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει επιφορτιστεί με αυτό το περίπλοκο ζήτημα Υπάρχει αυτή η ομάδα πυρογνωμόνων για τις ηθικές αξίες και θα ήθελα να προσθέσω ότι βεβαίως καλό είναι να υπάρχουν ηθικές και γραμμές αλλά δεν αρκεί ο ίδιος ο κλάδος, η διαβιομηχανία να αποφασίσει εάν θα ακολουθήσει αυτές τις αρχές ή όχι. Και αυτό που με τρομάζει είναι ότι για την ώρα ακούω συχνά ότι αυτό που θα γίνει εθελοντικά θα αποφασίσουν οι ίδιες επιχειρήσεις αν θα εγκρίνουν τις κρατικές γραμμές ή όχι. Δεν νομίζω να είναι αυτή η σωστή προσέγγιση για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανεξαρτησία, τις ελευθερίες. Αυτή είναι η δική μου προσωπική συνεισφορά στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ναι, έχω και σε μια άλλη συνάντηση να πάω, Πρόεδρε. Δυστυχώ δεν μπορώ να μείνω περισσότερο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο για συζήτηση. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις προς τους ομιλητές. Τώρα είναι η στιγμή για τις ερωτήσεις αυτές. Παρακαλώ να μας συστηθείτε, να μας πείτε προς ποιον απευθύνεται το ερώτημα και μετά να θέσετε το ερώτημά σας. Παρακαλώ εσείς κυρία. Ναι, καλό απόγευμα. Έχω μια μεγάλη εμπειρία και γνώση από διλήμματα ηθικής επιχειρήσεις ε, ιδιωτικές αλλά και στο δημόσιο τομέα. Μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ ποιον εκπροσωπείτε, από πού έρχεστε και σε ποιον απευθύνεστε. Ναι, συγγνώμη. Είμαι ο Άιβαν Μπιέφνο, συμμετέχω σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Ελεύθερης Σκέψης. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι τα τεχνικά σχέδια βάζουν την ηθική στο κέντρο, στο επίκεντρο και θέλω να, να ψυχαρώ την, ε, το Κοινοβούλιο για αυτήν την ε, προσέγγιση. Πολύ καλές αυτές οι αρχές, πρέπει όμως μετά να παρακολουθήσουμε τι γίνεται στην εφαρμογή, στην πράξη. Διότι έχω δει, έχω ακούσει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που λένε ότι κάποιοι από τους ε, εργαζόμενους τους είναι πεπαλαιωμένοι, είναι ξεπερασμένοι. Δεν ανταποκρίνονται στις ε, ε, απαιτήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης και πρέπει να αντικαταστηθούν από άλλους. Ξέρετε, πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα προστατευτικά. Πρέπει να υπάρξουν συστάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, διότι και αυτό έχει να κάνει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ένας άνθρωπος δεν είναι πεπαλαιωμένος. Μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να μιλάμε ότι είναι πεπαλαιωμένος. Αυτό. Μάλιστα. Θέλει κάποιος να αντιδράσει σε αυτό που μόλις υπόθηκε. Ε, καλό είναι να θέλετε πάντως ερωτήματα, κατά προτίμηση. Ναι, παρακαλώ. Ε, ναι, όλοι συμφωνούν με αυτό που λέτε. Πρέπει να γνωρίζουμε, να αντιληφθούμε ότι δεν δημιουργούμε εδώ έναν ιδανικό κόσμο όπου έχουμε τις υψηλότερες αρχές και τις μέγιστες. Προσπαθούμε απλώς στην εφαρμογή μας να είμαστε σωστοί. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να συστήσω όχι μόνο να θέσουμε όλες τις ηθικές αρχές, αλλά να σκεφτούμε ποιο θα είναι το περιβάλλον και το ευρωπαϊκό περιβάλλον αν θέλετε που είναι μεταξύ των Κινέζων ε, και την Silicon Valley ας πούμε ε, εφόσον λοιπόν ψάχνουμε ευρωπαϊκές λύσεις καλό είναι ε, να πληρούμε κάποιες προϋποθέσεις που προλέπει η παγκόσμια οικονομία και έχοντα αυτό κατά νου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Ε, thank you. Now, John this... Ο Τζον Χάουαρτ τώρα, ευρωβουλευτή, Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πάβελ. Δύο-τρία σύντομα σχόλια και ένα ερώτημα προ την Μπάρμπαρα Πριντσάκερ ε, που έκανε μια πολύ καλή παρουσίαση νωρίτερα ε, για τα ηθικά ζητήματα. σε σχέση με αυτό που είπε η Μάντι, είναι προφανές ότι η τεχνολογία ε, βεβαίως δημιουργεί κέρδος αλλά δημιουργεί και ε, μονοπόλια, δημιουργεί ανισότητες διότι αυτό ακριβώς συνέβη με όλες τις προηγούμενες φάσεις της τεχνολογικής προόδου γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ποιες είναι οι προκλήσεις ρύθμιση ε, σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, δίκαιο ανταγωνισμό βιώσιμη ε, και δίκαιη λειτουργία της αγοράς ε, Ιδάλλως δεν θα είναι δεν θα πάμε πουθενά. Τώρα, αυτοί που δημιουργούν την τεχνητή νοημοσύνη ε, είναι μία πάστας. Το να εισαγάγουμε διαφοροποίηση εκεί είναι περίπλοκο. Δεν είναι κάποιοι ε, ε, λευκοί άντρες ε, μεσαίας τάξης ε, που ακολουθούν αυτές τις αρχές ε, και αυτές τις προκαταλήψεις και αυτές τις αξίες. Αυτό είναι βασικό να μην συμβεί. Ίσως να θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτού, κυρία Πράιντσακ. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Το πρόβλημα της δημιουργίας της τεχνολογίας αυτής έχει να κάνει και με το όραμα των δημιουργών. Ε, ταυτόχρονα, ίσως να είμαι αισιόδοξη σήμερα, ε, δίνεται μεγάλη προσοχή αυτή τη στιγμή στα ζητήματα που αναφέρατε. Ότι δεν μπορούμε δηλαδή, να ρυθμίσουμε τον ανταγωνισμό δίκαια εάν επικεντρωθούμε στις επιπτώσεις για τους καταναλωτές μόνο σε επίπεδο τιμή. Διότι α, αυτά συμβαίνουν με την νομοθεσία antitrust. Ε, επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ακόμα χειρότερη από κάποιου κακού ανθρώπου ε, εάν δεν προσέξουμε είναι θέμα εταιρική ευθύνη αλλά και επιχειρηματική στρατηγική από του δημιουργού να αποδείξουν ότι έχουν λάβει υπόψη αυτέ τι ανησυχίε. Το λέω στου φοιτητέ μου σήμερα, αν γίνεται εμπειρογνώμονε στο μέλλον σε ζητήματα τεχνητή νοημοσύνη και ηθική, αυτή, αυτή η δουλειά ε, σίγουρα έχει μέλλον. Διότι αν κάποιος, ακόμα και κάποιο θεωρεί ότι δεν το χρειάζεται αυτό από ηθικής πλευρά, θα το χρειάζεται από πλευρά επιχειρηματική στρατηγική. Βεβαίω, εντάξει, άλλε μέρε είμαι πιο αισιόδοξη. Θεωρώ ότι έχουμε χάσει τη μάχη, α πούμε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ ο κύριο Τούνα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση. Ναι. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την Εσθονία στο Κοινοβούλιο αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ για τι συνεισφορέ σα. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και χρήσιμα αυτά που ακούσαμε. Να κάνω όμω και κάποια σχόλια. Μιλάτε για την αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται και με την ιερότητα. Το είπε και ο Ραβίνος. Η, η ζωή είναι ιερή. Και φοβάμαι ότι έχει χαθεί αυτός ο όρος, τον τρόπο σκέψη μας, τον καθημερινό και στην κρίση μας. Διότι τελικά τα πάντα γίνονται και τίποτα πια δεν είναι ιερό. Δηλαδή ε, η δράση μας είναι σε οριζόντιο επίπεδο μόνο. Επίση, συμφωνώ βεβαίω ότι καθήκον μα είναι να διαφυλάξουμε αυτόν τον κόσμο. ενέπνευσε η πρόταση να προωθήσουμε ε, την κλασική ε, ε, λογοτεχνία και βιβλιογραφία αναφερθήκατε στη βίβλο, στο Σέξπιρ ήδη από τα δεκαετία 30 υπήρχε αυτή η εικόνα η, η εφιαλτική του μέλλοντος όπου ο κόσμος δεν ασχολείται πια με αυτά και διέπεται μόνο από την τεχνολογία χάσανε τον Σέξπιρ και τη βίβλο και όλη την κλασική λογοτεχνία η οποία, την οποία κρύβουμε και απαγορεύουμε. Νομίζω ότι και αυτά τα έκανε ο Χίτλερ, έτσι. Το θέμα λοιπόν είναι τι γίνεται στο κεφάλι του μέσου ανθρώπου που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και που όλο και πιο συχνά δεν έχει ανεξάρτητη κρίση και σκέψη ηθική. Και αυτό αφορά και τη δυνατότητα που έχει κάποιος να διαγράφει. Όταν διαγράφει κανείς κάτι, καταστρέφει. Διαγράφουμε λοιπόν ότι δεν μας αρέσει και δεν έχουμε ηθική κρίση. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να διαφυλάξουμε αυτόν τον κόσμο σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα να οθήσουμε τους πολίτες να είναι πιο ανεξάρτητοι ή οι ανεξάρτητοι πολίτες να έρθουν στο προσκήνιο. Διότι οι πολίτες μας είναι όλο και πιο εξαρτώμενοι από το κράτος, από τις εταιρείε, από το διαδίκτυο. Είναι εξαρτώμενοι λοιπόν, δεν είναι ανεξάρτητοι σε ό,τι αφορά την ηθική τους κρίση. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ξεκινώντας από την κλασική παιδεία. Any reaction Κάποιος άλλος παρακαλώ, ο Ραβίνος. σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επισημάνεται τον όρο ιερός που ανέφερα και εγώ και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, σε αυτήν την Ήπειρο έλαβε χώρα το ολοκαύτωμα. Ε, οι άνθρωποι έχασαν την επαφή με το ιερό της ζωής και μας τρομάζει το ότι βλέπουμε κηρύγματα μίσους ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρχαν οι ε, ε, δεχθέστατες τρομοκρατικές πράξεις μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και ως κοινωνίες πρέπει σήμερα ακόμα περισσότερο να εκτιμούμε την αξία της ζωής. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για την ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα συμπεριέλαβε έλαβε ε, ε, αρχηγούς ομολογιών ε, γιατί η πίστη έχει πάρα πολλά να συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται γιατί η ιερή φύση της ζωής πρέπει να είναι καθοριστική σημασία για όλες τις μελλοντικέ σκέψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Η κυρία παρακαλώ. Είμαι η Σουζάννα Ντράγκομπιρ, είμαι ε, βοηθός στο Κοινοβούλιο, αλλά γράφω και το διδακτορικό μου και έχω κάποιες ερωτήσεις γιατί έχω και τις δικές μου ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί και ίσως μπορείτε να με βοηθήσετε. Μήπως είναι πολύ αργά για να ε, θεσπίσουμε κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη και για τις ε, ηθικές κατευθυντήριες γραμμές, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη ε, τροφοδοτείται από τα big data και η Ευρώπη δεν είναι ιδιοκτήτης των big data. Πώς μπορείτε να καταλήγετε σε μία λύση ενός εργαλείου το οποίο ε, ή να έχετε κατευθυντήριε γραμμέ σε διεθνέ επίπεδο, γιατί τελικά οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα είναι εκείνε που έχουν τα big data και που ε, φτιάχνουν την τεχνητή νοημοσύνη. Εμεί είμαστε ε, πολύ πίσω οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν έχουν την αρμοδιότητα για να επιβάλλουν οτιδήποτε στην Κίνα, παραδείγματο χάρη. Άρα, γεωπολιτικά έχουν το δικαίωμα να κατασκευάζουν στρατιωτικά ρομπότ. Ίσως ε, μπορείτε να μου απαντήσετε και σε αυτό πέρα από τις ηθικές επιφυλάξεις ε, και τα γεωπολιτικά στοιχεία. Θέλει κάποιος από εσά να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Θα κάνω ένα σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία δύο χρόνια ε, τα έχω περάσει μελετώντας την παραπλάνηση και τη διασπορά ψευδών δύσεων και τους τελευταίους ε, έξι μήνες ασχολούμαι με την τεχνητή νομοσύνη. Αλλάζουν πάρα πολλά. Η ηθική της τεχνητής ε, νομοσύνης τα τελευταία χρόνια είχαμε ένα έγγραφο σχετικά με την, το σχεδιασμό της ηθικής. Επίσης το Ενωμένο Βασίλειο ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Το Νοέμβρη είχαμε τη δήλωση του Μόντρελ για την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε και εσείς ε, τη δική σας ε, ομάδα υψηλού επίπεδου. Ξέρετε, για τους απλούς ανθρώπους δημιουργεί σύγχυση το να υπάρχουν όλα αυτά που να τρέχουν παράλληλα. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι νόημα έχουν όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω αν έχετε εσείς ένα σχόλιο ως Προεδρείο για το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερο ε, συντονισμό ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές πρωτοβουλίες. Γιατί τα πράγματα προχωράνε πολύ γρήγορα και δημιουργούν σύγχυση στους ανθρώπους. Ε, τελικά, ε, τις κατευθυντήριες γραμμές ποιον λαμβάνουμε υπόψη μας. Και όσον αφορά ε, τη διασπορά ψευδών λίστεων, 130 βιβλία έχουν δημοσιευθεί. Και αν προσπαθεί κανείς ε, να ε, είναι ενημερωμένος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά είναι απλώς μια έκκληση από εμάς. Θα καταγράψουμε την ερώτηση. Ευτυχώς, δεν ξέρω, εσείς θέλετε να απαντήσετε. Ε, ξεπερνάω τις αρμοδιότητές μου, αλλά θέλω να σας πω ότι πρόσφατα ακούσαμε σε συζητήσεις στο ε, Συμβούλιο της Ευρώπης στη Φινλανδία. Εκεί ακούσαμε ότι ένα διεθνές πλαίσιο θα μπορούσε να εξετάσει ε, την τεχνική πλευρά του διεθνού συστήματος αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ότι εκεί ε, πρέπει να υπάρχουν κάποια παγκόσμια εργαλεία γιατί αλλιώς ε, τα κενά ε, θα παραμείνουν και οι άνθρωποι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα κάνουν τη δουλειά τους. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κάπου ανάμεσα στην ηθική και τον νόμο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ο επαγγελματισμός. Δηλαδή υπάρχουν ειδικέ αρμοδιότητες, ε, υπάρχουν ε, οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Όπως και σε άλλους τομείς αναγνωρίζουμε τη σημασία των επαγγελμάτων. Ε, οι άνθρωποι λένε ότι εγώ τάσομαι υπέρ του ανθρώπινου καλού και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το στηρίξουμε μαζί με το ηθικό και το νομικό στοιχείο. Πρέπει να εξετάσουμε ε, και τα κίνητρα των ανθρώπων. Νομίζω ότι ε, κάνατε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να την απαντήσουμε. Δεν έχω βέβαια μια τέλεια απάντηση. Επισημάνατε ότι ε, το κλειδί είναι να έχει κανείς τα δεδομένα. Και όλοι μιλάμε ε, για αυτά τα δεδομένα, αλλά υποτίθεται ότι τα δεδομένα μπορούμε όπως και το πετρέλαιο να τα βγάλουμε από τη γη και να τα διηλύσουμε δεν είμαστε ιδιαίτερα συνεπείς με την έννοια ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την πρόσβαση στα δεδομένα ως ε, ένα νέο στοιχείο της νομοθεσίας ε, κατά των ε, ομίλων επιχειρήσεων. Κάπως το χάνουμε αυτό απολύτως και Διαφωνώ απόλυτα με τον Πίτερ. Θεωρώ ότι η ε, κυριαρχία των data χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις και τους εκπροσώπους λόμπι για να δημιουργήσουν ένα ειδικό καθεστώς ιδιοκτησίας όπου θα λένε στους ανθρώπους θα, θα μας δώσεις ε, τα δεδομένα, θα σε πληρώσουμε και δεν θα υπάρχει ε, καμία συλλογική ευθύνη. Δεν λέω ότι το κάνουν όλοι αυτό, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και το πρόβλημα που θέσατε είναι πραγματικά το κέριο πρόβλημα στην ε, τεχνητή νοημοσύνη. Δυστυχώς, λέει ο Πρόεδρος, ε, δεν έχουμε πλέον χρόνο. Έχουμε εξαντλήσει το χρόνο για αυτό το πρώτο πάνελ. Έτσι, κυρία Αντιπρόεδρε, ε, θα ήθελα να σας δώσω τώρα την διεύθυνση της συζήτησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, συνάδελφο για αυτό το πρώτο πάνελ. Ε, θα μιλήσω και εγώ σύντομα, γιατί η κυρία Καϊλή θα προεδρεύσει ε, στο επόμενο πάνελ. Εγώ θα επιτρέψω άλλο ένα σχόλιο, αν θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Είμαι ο πατήρ Γεώργιος Λέκας, που εκπροσωπώ την Εκκλησία της Ελλάδας. εξοχότατη. Νομίζω ότι σήμερα για μας είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να συζητήσουμε το σχέδιο ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την τεχνητή νομοσύνη. Κάτι που μόλις δημοσιεύτηκε. Το δικό μας το γραφείο αναγνωρίζει αυτή η συζήτηση ω ένα απαραίτητο βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου όμω να παραθέσω από άλλε κατευθυντήριε γραμμέ για την τεχνητή νομοσύνη που εκπονήθηκαν το 18 από το Συμβούλιο τη Ευρώπη και παραθέτω θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη αντίληψη, μια αντίληψη που εξετάζει όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, αλλά και τη λειτουργία των δημοκρατικών και κοινωνικές και ηθικές αξίες. Τέλος της παράθεσης. Η ε, βασική μας κριτική κατά των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αυτές ε, δεν λαμβάνουν υπόψη του τι ευρωπαϊκέ ηθικέ και κοινωνικέ αξίε. Δεν τι λαμβάνουν καθόλου υπόψη του. Και μετά. πώ μπορούμε στην Ευρώπη να έχουμε αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν λαμβάνουν υπόψη οι ηθικέ και κοινωνικέ αξίε. Οι ευρωπαϊκέ ε, ηθικέ αξίε, όπω η ευθύνη, η ε, άφεση αμαρτιών, η εμπάθεια, συγγνώμη, η κατανόηση, αυτά θεωρούνται ως ε, στοιχεία που δεν είναι αυτόνομα, που τελικά δεν είναι και το σημείο κίνηση τη Επιστημονική Επιτροπή που, κατέγραψε, που συνέταξε αυτό το έγγραφο. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτόνομος, αλλά επηρεάζεται από κοινωνικές επιδράσεις και μπορεί να ευημερίσει μόνο με την αγάπη των υπόλοιπων συνανθρώπων. Για αυτούς του λόγους πιστεύουμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα και να προάγουμε τις ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες. Όχι να βάλουμε όρια στην αυτονομία των ανθρώπων, αλλά για να τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να ζουν μια ζωή με νόημα με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες. Πρόεδρος, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η παρέμβασή σας. Αυτά που θέλετε να πείτε τα δώσαμε στους συναδέλφους. Συστήνω σε όλους να τις διαβάσουν. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν ε, θα δώσω το λόγο ε, στον κύριο καθηγητή ε, για να τοποθετηθεί. Ίσως μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ λιγάκι σε αυτό που μόλις ελέγχθη. Η αυτονομία και η κατανόηση του ανθρώπου αυτό μας επαναφέρει στη δική σας τη θέση, Μπάρμπαρα, εδώ δύο σχόλια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλες οι έννοιες μπορούν να είναι αντικείμενο κατάχρησης, ακόμα και η νομοθεσία για τους ομίλους επιχειρήσεων. Ε, όλα μπορούν να είναι αντικείμενο καταχρήσεων. Και εγώ προσωπικά θεωρώ την κυριαρχία των δεδομένων ως κάτι το οποίο μπορεί κανείς να ελέγξει και όχι να οικειοποιηθεί. Γιατί συμφωνώ η έννοια της ιδιοκτησίας, όπως αναφέρετε και εσείς την αλληγορία αυτή με το πετρέλαιο, αυτό τελικά δεν θα κατορθώσει να ε, κυριαρχήσει σε ένα κόσμο που θα καθοδηγείται από την τεχνητή νομοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν την ερμηνεία της αυτονομίας πρέπει να την ε, ταυτίζουμε και με τον έλεγχο και με οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει τον έλεγχο του ε, ατόμου. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι δηλαδή να δίνει κανείς καταρχήν τη συνένεσή του και μετά να χάνει πλήρως την αυτονομία. Γι' αυτό επανέρχομαι στη δική σας την ερώτηση ε, της ε, κυρίας που κάνει διατριβή και εδώ θέλω να σας απαντήσω ότι σε αυτή την ομάδα των ε, θρησκευτικών αρχηγών ο ένας Βρετανός φιλόσοφος δημοσίευσε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Χωρίς αισιοδοξία». Και νομίζω ότι βλέποντας τι διαδραματίζεται, πράγματι δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Συμφωνώ μαζί σας ότι η απεσιοδοξία μας έχει κατακυριεύσει. Όμως ε, τελικά υπάρχουν κάποια υπερβατικά συστήματα πίστης και εμείς ε, πρέπει να αντισταθούμε για να διατηρήσουμε την αυτονομία μας πάση θυσία για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια η οποία αφενός εντάσσεται στις σχέσεις αλλά ε, ο τελικός στόχος είναι η αυτονομία. Και αν ε, έχετε απόψεις που να αφορούν ας πούμε ε, τις, ε, τους ομίλους επιχειρήσεων και τη σχετική νομοθεσία όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο μπορείτε αυτές απόψεις να τις εκφράζετε αλλά μην ξεχνάτε παρακαλώ ότι υπάρχει αυτή η ένταση και έχουμε εγκλωβιστεί ανάμεσα στην ένταση αφενός του Silicon Valley και αφετέλου προσεγγίσεων περί κρατικού καπιταλισμού. Αν δεν μπορέσουμε να ανέλθουμε σε αυτό το επίπεδο, θα αποτύχουμε. Τελευταίο σχόλιο και μετά θα περάσουμε στο επόμενο πάνελ. Ναι, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Δύο φράσεις. Κάποιος εδώ είπε ότι πρέπει να βασιστούμε στην συνείδηση των ανθρώπων να κάνουν επιλογές. Έχει λοιπόν κάποιος από εμά την επιλογή αυτήν. Δεύτερον, ε, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες και των ιατρών ε, υπάρχει ένας κίνδυνος με ό,τι αφορά το G4. Πρόσφατα ε, έλαβα και μια έκθεση για το G5 που θα προκύψει στην Ευρώπη και στην, Βέλγιο. Ε, μήπως τελικά πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ. Okay, questioning choice. Which... Μάλιστα. Το θέμα της επιλογής, κατά πόσο υπάρχει όντω επιλογή. Θέλει κάποιος να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν βλέπω να με κοιτάζει κανεί. Θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς, κυρία μου, για την επιλογή. Μετά ενδιαφέρον και το ερώτημα για την ηθική που δεν αρκεί και που χρειάζεται και νομοθεσία. Συγγνώμη που σας βάζω στην πρώτη γραμμή. Νομίζω ότι έχω ήδη πει πολλά, έχω μιλήσει πολύ. Ε. Θα μπορούσα να, δώσω, να αφήσω το λόγο και σε κάποιον άλλον, εν περιπτώσει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε για τη, συμφωνή, τη σημασία της επιλογής, της δυνατότητα επιλογής και θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι όταν μιλάμε για ρύθμιση με την ευρύτερη έννοια τη τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύνολο των πολιτικών παρεμβάσεων είναι στη διάθεσή μας. Δεν είναι μόνο είτε ηθική, ηθικές αρχές, είτε νομοθεσία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πάντα. Όλα αυτά. Ορισμένε φορές και η κατάλληλη επιλογή της ορολογίας είναι κρίσιμη. Νομίζω ότι συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε ε, την τεχνολογία. Και πρέπει αυτό να το λέμε. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε, να ελέγξουμε αυτό το κλάδο. Σας ευχαριστώ όλους που συνεισφέρατε σε αυτή την εξαιρετική συζήτηση. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά ε, θα δώσω τη σκητάλη στην φίλη και συνάδελφο την κυρία Καηλή. Έτσι θα μπορέσω να παρακολουθήσω εγώ τη συζήτηση χωρίς να εργάζομαι. Προσχολείται με την, είναι επικεφαλής μάλλον της Επιτροπής ΣΤΟΑ. Συμμετείχα στην Επιτροπή αυτή που κάνει πολύ καλή δουλειά και πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρία Καηλή